ολοκληρωθεί ε, η ημερήσια διάταξη ό,τι αφορά τις συζητήσεις μας. Για σήμερα περνάμε στην ψηφοφορία αυτών των ε, ψηφισμάτων. Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση σε ό,τι αφορά τις ε, μεταδοτικές ζωνόσους. Θα το περιλάβουμε στα πρακτικά